Uh, uh, λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει κατά ένα τέταρτο, λίγο πάνω από ένα τέταρτο, την ε, έναρξη της συνεδρίασής μας. Γι' αυτό ας αρχίσουμε με την εργασία μας. Είμαστε τώρα στο σημείο 23, η πρόοδος των τριμερών διαπραγματεύσεων. Όπως γνωρίζετε, πριν από τις ε, καλοκαιρινές διακοπές καταλήξαμε σε μία συμβιβαστική ε, συμφωνία με το Συμβούλιο σε μία δέσμοι σεμάτων, προτιμησιακές συμφωνίες, Πακιστάν και άλλα θέματα. Καταλήξαμε λοιπόν σε συμφωνία με το Συμβούλιο και όλα αυτά τα ντοσιέ πλέον τα έχουμε συμφωνήσει με το Συμβούλιο. Αλλά υπάρχουν δύο σημαντικές εξαιρέσεις. Υπάρχει και μία παγωμένη πρωτοβουλία ε, στο, στο, στα ράφια του Συμβουλίου και το άλλο είναι το Omnibus. Και αρχίζω λίγο και ανησυχώ για αυτούς τους δύο φακέλους. the end of this Για το Omnibus λοιπόν και το Omnibus 2 ε, δεν ξέρω το Συμβούλιο γιατί κολλησιεργεί θα πρέπει να προσαρμοστεί το νομοθετικό εκτιμένο στις απαιτήσει ε, της συνθήκης της Λισαβόνας και των εφαρμοστικών πράξεων. Δεν πρέπει λοιπόν να κολλησιεργούμε σε αυτούς τους δύο φακέλους. Γι' αυτό θα προτείνω στην επόμενη συνάντησή μας με το Συμβούλιο μια πάρα πολύ σκληρή θέση. Ή είτε το Συμβούλιο θα απαντήσει στις θέσεις μας για το όμνιμπους που θα μας επιτρέψει την έναρξη των διαπραγματεύσεων ή κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εφαρμόσουμε αντίπεινα στη θέση του Συμβουλίου. Είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά του Συμβουλίου. Το άλλο θέμα είναι η μακροοικονομική βοήθεια σε διάφορες χώρες, στη Μολδαβία αν δεν κάνω λάθος ε, και Γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν και πάλι το Συμβούλιο να προτείνει κάτι λογικό μέσω της ε, διαδικασίας επιτροπολογίας. Δεν μπορούμε να εξαρτώμεσα από την ε, αλλαγή διαθέσεων του Συμβουλίου ή τις, ε, τις δυσκολίες που μας φέρνουν. Λοιπόν, θα ε, δείξω την ε, νευρικότητα που έχουμε τώρα, την ανησυχία που έχουμε για αυτούς τους φακέλους. Και εάν δεν σημειωθεί πρόοδος σε αυτούς τους δύο φακέλους από πλευρά Συμβουλίου, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια πολύ σκληρή θέση. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους απειλήσουμε. να τους απειλήσουμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με το Συμβούλιο σε άλλα θέματα, σε άλλους φακέλους που τους ενδιαφέρουν πολύ. Παραδείγματο χάρη, η Καραϊβική και η Κεντρική Αμερική και οι, οι κανονισμοί διασφάλισης. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Μπερτ Λάγκερ, τον εισηγητή ε, που είναι ο ε, εισηγητής για, τις, ε, για τους κανονισμούς διασφάλισης. Αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο θα συζητήσουμε με το, φάκελο με την Κεντρική Αμερική και των άλλων για το Περού έχουμε ε, διατυπώσει ένα σωρό αιτήματα από πλευράς Κοινοβουλίου για να ε, εξασφαλίσουμε ένα δίκτυο προστασίας ε, των προϊόντων επίσης για την υποχρέωση εποπτείας, παρακολούθησης και για την σωστή συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαδικασίες. Το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει μια άκαμπτη στάση και δεν δέχεται ούτε καν αυτά τα οποία είχε δεχθεί στους κανονισμούς διασφάλισης με την Νότιο Κορέα. Ε, εάν δεν καταλήξουμε συμφωνία, αύριο θα χρειαστούμε και περαιτέρω γύρους διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, πρέπει να συμφωνήσουμε επιτέλους, αλλά τουλάχιστον να έχουμε και μία εναλλακτική λύση για μία συμφωνία που θα επιτευχθεί αργότερα, αν δεν γίνει αύριο. Ο, το Συμβούλιο ήρθε σε επαφή μαζί μου για διαδικαστικά θέματα και αύριο θα πρέπει να υιοθετήσουμε το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία. Συνήθως στον πρώτο γύρο του, διαλόγου, του τριλόγου των τριμερών διαπραγματεύσεων γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων και συμφωνούμε στα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία στις τριμερείς διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ, Μπερτ Λάγκε. Άλλα σχόλια για αυτό το θέμα. Όχι, ωραία. Τώρα, στον κανονισμό πρόσβασης αγοράς που ψηφίστηκε στο Στρασβούργο. Έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τώρα την πολιτική απόφαση. Αυτό το ολοκληρώσαμε και γι' αυτό αναμένουμε την επόμενη κίνηση του Συμβουλίου. για να μπορέσουμε αργότερα να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο. 24. Δραστηριότητες εποπτικής ομάδας. Ε, εδώ υπάρχουν διάφορα, διάφοροι τομείς ως εισηγητής που είμαι εγώ για την μόνιμη εποπτική ομάδα με τις Ηνωμένε Πολιτείες, πρέπει να πω ότι αυτή η εποπτική ομάδα ήταν πολύ ενεργή, οργανώσαμε μία συνάντηση με τους Ευρωπαίους συμβαλόμενους και εκεί εκπροσωπήθηκαν όλοι οι τομείς ε, της Ευρωπαϊκής ε, των ευρωπαϊκών κλάδων και καταγράψαμε τις θέσεις τους για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένε Πολιτείε, όπως είπαμε. Και η συζήτηση ήταν πολύ ζωηρή. Ένας, ένας, ε, συμβαλο, ένας ενδιαφερόμενος, ένα μέρος των συμβαλωμένων έδειξε λιγότερο ενδιαφέρον, αλλά όλοι οι άλλοι περίπου ε, θα έλεγα ότι ήταν ενθουσιώδης για την ιδέα αυτή της έναρξης των, των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Στρασβούργο όχι. με τον πρέσβη με την πρέσβη Μίριαμ Σαπίρο. η οποία είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις με την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή, την συνόδεψε ο Βίλιαμ Κανάρ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, των στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Συζητήσαμε τη δική μου, το δικό μου σχέδιο γνωμοδότησης και ε, σχολιάστηκε γενικά ε, ο στόχος όμως της συνάντησης ήταν, ο σκοπός μάλλον, ήταν να ακούσουμε τις δικές τους απόψεις. Για την Ιαπωνία δεν βλέπω τον Μάρτιν Καζάκ να είναι εδώ, αλλά από ό,τι ξέρω από τις σημειώσεις της γραμματείας έγινε μία συνάντηση με επιχειρηματίες και επιχειρηματικές οργανώσεις και επειδή είμαι σκιώδης εισηγητής για την Ιαπωνία, και εγώ παρόν. Δεν μπόρεσα να μείνω μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Δεν ήταν και πολύ μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων τότε, αλλά ήταν μια χρήσιμη συνάντηση. Και εκφράστηκαν διάφορες απόψεις, διαφορετικές απόψεις. Ορισμένοι είχαν την άποψη ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις πριν, ε, προτού έχουμε την πολύ ισχυρή δέσμευση της Ιαπωνικής πλευράς. Άλλοι ήθελαν να μπουν περισσότερα θέματα στο διαπραγματευτικό τραπέζι και να πιέσουμε τους Ιάπωνες. Και πρέπει να πω ότι τουλάχιστον στις δύο αυτές περιπτώσεις οι εποπτικές ομάδες ε, έδειξαν ότι επιτελούν ένα καλό έργο, επιβεβαίωσαν δηλαδή την αξία τους, ε, της εργασίας τους και κατά κάποιο τρόπο αποκεντρώνονται και οι εργασίες της Επιτροπής μας. Επιμένω όμως ότι αυτές οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές και προσβάσιμες για όλα τα μέλη της Επιτροπής. Δεν, είναι, δεν υπάρχει τίποτα το κρυφό ή μυστικό και όλα τα μέλη μας ε, είναι ευπρόσδεκτα σε αυτές τις συναντήσεις των υποπτικών ομάδων. Σχόλια παρακαλώ, παρατηρήσεις. Όχι. Επόμενο θέμα είναι το 25. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδάς αναφορά τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε αυτή τη διαδικασία συνένεσης. Είμαστε η επί της ουσίας επιτροπή, ο εισηγητής μας είναι ο Πίτερ Στάσνη, ο οποίος είναι και ο εισηγητής για τις σχέσεις μας με τον Καναδά και του δίνω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια σας, για την εποπτική ομάδα ως ε, συμμετέχονται εισηγείται για τον Καναδά. Θα συναντηθούμε αυτή την εβδομάδα. Ήταν μάλλον να συναντηθούμε αυτή την εβδομάδα, αλλά το αναβάλαμε για την επόμενη, διότι γίνονται διάφορε εσωτερικέ διαπραγματεύσει. Είμαστε λοιπόν καλύτερα ενημερωμένοι και έχουμε ήδη ορίσει χώρο και χρόνο. Έτσι θα είμαστε σε καλύτερη θέση να μπορέσουμε να είμαστε καταλέμενοι ενημερωμένοι και για τις μελλοντικέ μας συναντήσεις τώρα. Όσον αφορά την τελωνιακή συνεργασία και τα θέματα ασφαλείας και τελωνίων και τη διαχείριση κινδύνων, αυτό ουσιαστικά συνίσταται σε προσθήκες και σε επέκταση της συμφωνίας, της αρχικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά το 1998. Στη συνέχεια ο Καναδάς αποφάσισε να επεκτείνει αυτή τη Συμφωνία Τελωνικής Συνεργασίας το 2005 ζήτησε επέκταση και παράταση. Το 2009, αν δεν κάνω λάθος, το Συμβούλιο έδωσε την εντολή στην Κομισιόν και το 2011 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Βασικά η κατάσταση σε μένα φάνηκε λίγο περίεργη διότι είχαμε την πρώτη ανάγνωση και μετά από περίπου έξι μέρες Υποτίθεται ότι θα έχουμε την έγκριση του Συμβουλίου και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου πριν καν προλάβουμε να ολοκληρώσουμε εδώ και ανεξαρτήτως τι θα γίνει στο Κοινοβούλιο θα συμφωνηθεί. Πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία όπου το Κοινοβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο. Ε, δεν χρειάζεται να βιαστούμε Εμείς θα έχουμε τον τελικό λόγο έγκρισης ή έγκριση νέα συμφωνία συμφωνια ελληνικής συνεργασίας και αμοιβαίας αρρωγής ε, θα πρέπει να επεκταθεί στη διαχείριση κινδύνων της αλυσίδας εφοδιασμούς. Ε, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, όπω είπα, ξεκίνησε το 1998 σε αυτόν τον τομέα και οι πόρτε είναι ανοιχτέ. Έχουμε καλέσει του διαφορού ενδιαφερομένου. Προ το παρόν δεν αντιμετωπίζω καμία δυσκολία. Οπότε ολοκληρώνω εδώ και αν κάποιο θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο ή κάποια ερώτηση, ευχαρίστω θα την απαντήσω. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε για την παρουσία σα. Το σχέδιο αποφάσεως του Συμβουλίου βρίσκεται στα χέρια σας. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Αργότερα ο εισηγητής ε, θα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης σύμφωνα με τις σημειώσει μου. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 24 Σεπτεμβρίου για τη μετάφραση και εξέταση μάλλον της, ε, του σχεδίου έκθεσης θα λάβει χώρα στις 10 και 11 Οκτωβρίου εδώ στη συνεδριάση μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις συζητήσεις την πρώτη παρατήρηση να κάνει η κυρία Σελβάνα Κοχμέριν. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη, απλά ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις παρατηρήσεις του και την αξιολόγησή του αυτή της απόφαση του Συμβουλίου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Θεωρώ ότι δεν προβλέπεται να υπάρξουν ιδιαίτερε διαφωνίες όσον αφορά το περιεχόμενο. Πρόκειται για μια προσ... κάτι συμπληρωματικό προς την Συμφωνία ΣΥΤΑ και είναι... Πρόκειται για μια διεύρυνση ουσιαστικά τη συμφωνία σε άλλου τομεί. Ωστόσο, συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε. Ω Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μεριμνήσουμε ώστε οι κανόνε μα να τηρούνται και να διαδραματίσουμε το ρόλο που μα παρέχουν οι συνθήκε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό όντω θα λάβει χώρα και ότι οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι στο ευρωπαϊκό σκηνικό θα είναι ενημερωμένοι και θα όσο και εμεί Ευχαριστούμε πολύ για το έργο σα και ανυπομονούμε για περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστούμε, δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Α ζητήσουμε λοιπόν την άψη τη Επιτροπή, Κυρία Λίλιαν, σνίφτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ο κύριος Λίνιαν Προέρχομαι από την Digitaxus, επιφορτισμένη με τον συντονισμό των φορολογικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την παρουσίαση αυτής ε, της, και την εισαγωγή σε αυτή τη συζήτηση. Απλά ήθελα να προσθέσω δύο παρατηρήσεις όσον αφορά την παρουσίαση αυτού του σχεδίου απόφασης, της πρότασης απόφασης. Πράγματι, όπως ε, επισημάνθηκε από τον εισηγητή, το σχέδιο συμφωνίας για την ασφάλεια τη της αλυσίδας εφοδιασμού αποσκόπη στο να επεκτείνει στον τολωνιακό τομέα την τρέχουσα συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά. Μία επέκταση ουσιαστικά μιας αρχικής ε, συμφωνίας του 1998. Κατά τα τελευταία λοιπόν 15 χρόνια συνέβησαν πολλά. Αναδύθηκαν οι ανησυχίε ασφάλεια τη αλυσίδα εφοδιασμού ω μείζον θέμα ανησυχίε για τι τελωνιακέ αρχέ. Αναπτύχθηκαν νέα εργαλεία που επιτρέπουν στα τελωνία μέσω της χρήσης εργαλείων πληροφορική, να προσδιορίζουν καλύτερα τους κινδύνους, διευκολύνοντας ταυτόχρονα το εμπόριο. Αυτή είναι η προσέγγιση που υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολλά επίπεδα, διαχείριση κινδυνού πολλών επιπέδων. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι αποδεκτή και στον Καναδά. Έχουμε και αποδεκτικά στοιχεία γι' αυτό. Με την εκπόνηση του σχεδίου απόφασης που βλέπουμε σήμερα, ο σκοπός είναι οι τελωνιακές αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά να μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού που καθίσταται δυνατή με τα νέα εργαλεία και όπου είναι απαραίτητο χάρη στην ανάλυση των νέων απειλών για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα πω δύο γρήγορα λόγια για το εύρος της συνεργασίας που περιγραφτεί στο άρθρο 2 και πιο λεπτομερώς στο άρθρο 4 του σχεδίου απόφασης. Περιλαμβάνει για παράδειγμα την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων για τεχνικές διαχείρισης κινδύνων, την καθιέρωση αμοιβαίας αναγνώρισης σε πολλούς τομείς, αμοιβαία αναγνώριση τεχνικών διαχείρισης κινδύνων, προτύπων κινδύνων, ελέγχων ασφαλείας και προγραμμάτων ε, εμπορικής ε, συναλλαγής. Επίσης, περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με την επιφύλαξη της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και βάσει των απαιτήσεων προστασίας των δεδομένων. Επίσης περιλαμβάνει την καθιέρωση σημείων επαφής και διαπαφών για την ανταλλαγή δεδομένων, συνεργασία για τις επιθεωρήσεις και συνεργασία σε πολυμερή φόρα. Και ένα από αυτά τα σημαντικά πολυμερή φόρα είναι ο Παγκόσμιος Τελωνιακός Οργανισμός εδώ στις Βρυξέλλες. Από αυτές τις συνεργατικές δράσεις θα ήθελα να επισημανω που εμείς αναμένουμε ότι θα αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα αμέσως μετά από την υιοθέτηση της συμφωνίας. Πρόκειται για την αμοιβαία αναγνώριση των προγραμμάτων εμπορικής συνεργασίας, εμπορικής εταιρικής σχέσης. Ε, αντιστοιχεί σε ένα καναδικό πρόγραμμα που λέγεται Partners in Protection. το PIP δηλαδή. Πρόκειται, όπως είπα, για δράση που θα έχει πρώτη προτεραιότητα. Μετά από τις κοινέ προσπάθειες με τον Καναδά θα ακολουθήσουν συμφωνίες όπως αυτές που υιοθετήσαμε με την Ιαπωνία πέρυσι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα φέτος. η νομοθεσία για εξουσιοδετωμένο χειριστή που έχει καθιερωθεί εδώ και πέντε χρόνια είναι επιτυχής με τους Ευρωπαίους, ε, με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πάνω από 5.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ήδη πιστοποιηθεί, έχουν διαπιστευθεί είτε χάρη στη συμμόρφωσή τους με τους τελωνιακούς κανόνες, καθώς και φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή έχουν τα σχετικά πιστοποιητικά Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε επειδή πληρούν απαιτήσεις, υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι το δεύτερο πιστοποιητικό, αντιστοιχεί στο δεύτερο πιστοποιητικό που ε, αποτελεί κομμάτι τη αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ εταίρων. Οι ελπίδε μα λοιπόν είναι πολλέ ότι θα γίνουν περαιτέρω προσπάθειε για αμοιβαία αναγνώριση και θα φέρουν αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι οι συζητήσει μα με τον Καναδά θα πρέπει να εστιαστούν σε αυτό το συγκεκριμένο πρόθεσμο σχέδιο μόλις υιοθετηθεί η συμφωνία. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας, αγαπητοί συνάδελφοι, για οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συναδελφ, τη συναδελφό μου Κοχμαρέν για την συμμετοχή της. Αυτό βοηθάει να συμπληρώσουμε την συνεργασία μας για μια ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά. Εκτιμάμε ιδιαίτερα τι παρατηρήσει τη Κομισιόν και ανυπομονώ να καταλήξουμε και στο, σε ένα τελικό ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Το επόμενο βήμα μελέτη του σχεδίου έκθεσης στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Σημείο 26. Πρόκειται για την ίδια διαδικασία συνένεσης που αφορά μια διεθνή συμφωνία. Πρόκειται για την τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλων 1 και 2 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και του κράτους του Ισραήλ αφετέρου. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ΑΚΑ που συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ τεχνικό θέμα. Γι' αυτό αποφάσισα να ακολουθήσουμε απλοποιημένη διαδικασία και παρουσίασα το σχέδιο σύστασης ώστε να συνενέσουμε στην τροποποίηση αυτή της τεχνικής αυτής συμφωνίας. Κατά συνέπεια, και εφόσον πρόκειται για κάτι τεχνικό, παρακαλώ την Επιτροπή αν θέλει να μας πει κάτι. Ποιος εκπροσωπεί την Κομισιόν, παρακαλώ. Η κυρία Ντόρμα Μαρίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή. Και σωστά, όπως είπατε, πρόκειται για ένα πάρα πολύ τεχνικό φάκελο. Κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης και διαπραγμάτευσης μιας ε, συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ το 2010 υπήρξε ένα τεχνικό σφάλμα και το έγγραφο που έχετε απλώς στοχεύει στην διόρθωση αυτού του σφάλματος. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σας απασχολήσει περαιτέρω. Αρκετά χρόνο αναλώσαμε. Ευχαριστούμε την εκθεσή σας. Υπάρχει καμία παρατήρηση? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συνενέσουμε. Θα πρέπει να στείλουμε γι' αυτό το τεχνικό σφάλμα ένα ισχυρό μήνυμα στο Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε κατά τη συνένεση. Πρόκειται για κότι το τεχνικό, αλλά γιατί. Πρώτα απ' όλα, ε, να είναι τα πράγματα έτσι ως έχουν. Δεν με αφορά τόσο αυτή η συμφωνία, αλλά το γεγονός ότι επιδεινώνονται όλο και περισσότερο οι Ισραήλ. Ξέρουμε ότι στην χώρα αυτή όλο και περισσότερα υπάρχουν παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίω κατά των παιδιών. Ξέρουμε ποια είναι τα θέματα που υπάρχουν στη χώρα αυτή, γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υποφεληθούμε αυτή τη ευκαιρία για να αρνηθούμε τη συνένεση. Ευχαριστώ. Όλοι ξέρουν τη θέση μου σε σχέση με οποιαδήποτε βελτίωση των σχεσιών αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα με οδηγήσει αυτό και στο να απορρίψω μια ε, τεχνική τροπολογία, τεχνικού περιεχομένου τροπολογία για αυτό το θέμα. Είναι τεχνικού περιεχομένου, όπως ξέρετε. Πιστεύω λοιπόν ότι αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορεί η σύστασή μου να γίνει αποδεκτή. 19 Σεπτεμβρίου κατάθεση τροπολογιών, Οκτώβριο συζήτηση στην Επιτροπή, ε, Ολομέλεια του Νοεμβρίου συζήτηση στην Ολομέλεια. Τώρα, που είναι ο Αγλέμ Ντεζίρ, θα έχουμε μία κοινή συζήτηση για δύο θέματα για την εταιρική κοινωνική ευθύνα ευθύνη. Πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων για τις δύο αυτές εκθέσεις. Η πρώτη είναι γνωμοδότηση για την ε, Επιτροπή Επασχόλησης που είναι υπεύθυνη επί της ουσίας και η άλλη επίσης γνωμοδότηση για την Νομική Επιτροπή που είναι Υπεύθυνη επί της ουσίας. Οι εκθέσεις αυτές έχουν σχέση με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανανέωση της ε, στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 12-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και οι δύο επιτροπές, απασχόλησης και νομική, έχουν αποφασίσει να συντάξουν έκθεση πρωτοβουλίας και εμείς να συντάξουμε γνωμοδότηση. Παρά το γνωστό και για δύο διαφορετικές γνωμοδοτήσεις θα έχουμε ε, ενιαία ε, γνωμοδότηση. Δεν είναι εδώ Αρλέμ διότι ετοιμάζεται να αναλάβει νέες ευθύνες σε επίπεδο γαλλικής πολιτικής. Ετοιμάζεται να εκλεγεί Γενικός Γραμματέας Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας. Ζήτησε συγγνώμη για την απουσία του. Τον αντικαθιστά ο Μπέρτ Λάγκε. Μπέρντ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω το, να απολογηθώ για τον Αλάν Βεζίρ, Χαρλέμ Δεζίρ, δεδομένου ότι υπάρχει ένας νέος πρόεδρος της, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, στην ε, Φραγκφούρτη και γι' αυτό είναι πάρα πολύ αποσχολημένος εκεί. Εξ ονόματός του θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες του και είπατε ήδη ότι και οι δύο εκθέσει αναφέρονται σε μια ανακοίνωση της Κομισιόν για την ανανέωση της στρατηγικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και αυτή η ανακοίνωση είναι πραγματικά αξιοσημείωτη διότι ε, η, η προσέγγιση αυτή, η, η όλη θεωρία της εταιρική κοινωνικής ευθύνης έχει μετατραπεί, έχει αλλάξει. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη τέσκε περίπου πριν από 10 χρόνια στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε τρεις ανακοινώσεις της Κομισιόν, διάφορες ενέργειες έγιναν γύρω από αυτό το θέμα και όλα ο Αλέμ Ντεζίρ το 2010 παρουσίασε μία έκθεση ε, για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στο διεθνέ εμπόριο, στι διεθνεί εμπορικές συναλλαγές. Τώρα η προσοχή επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην προαιρετική συμμετοχή των εταιριών. Ε, ορισμένες εταιρείες έχουν υιοθετήσει διεθνή πρότυπα διεθνή standards, τα οποία αναφέρονται ε, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές ε, της, ε, του ΟΣΑ, η καινούργια πρωτοβουλία Nobel Compact, η... όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες διεθνείς και οργανισμοί που έχουν εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές ή γενικές, γενικούς προσανατολισμούς για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Όμως όλα αυτά είναι πολύ ασαφή και δεν είναι υποχρεωτικά, δεν υπάρχει καμία δέσμευση για αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές. Γι' αυτό θέλουμε η Κομισιόν να ζητήσει μεγαλύτερη δεσμευτικότητα, να ενισχυθεί το στοιχείο της δέσμευσης, έτσι ώστε να υπάρχει βεβαίως ε, μία μετατόπιση από το στοιχείο της εντελώς προαιρετικής και ασελούσιας συμμετοχής σε μία πιο δεσμευτική συμμετοχή, σε μία υποχρέωση ε, η οποία υποχρέωση επίσης θα, ε, θα αναγκάζει τις εταιρείε να σέβονται και τα διεθνή πρότυπα. Η, το ISO 26000 το πρότυπο ISO 26.000 θα μπορούσε να αποτελέσει το πρότυπο εκείνο που θα υποχρεώνει τις ε, διεθνείς εταιρείες ή μάλλον τις εταιρείες διεθνώς να κάνουν σεβαστές αυτές τις διατάξεις κοινωνικέ κοινωνικές Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Ε, πολλές εταιρείες έχουν ακολουθήσει τις ε, κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική ευθύνη ευρωπαϊκές εταιρείε. Πολλές όμως άλλες διεθνώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και ούτε θέλουν. Αυτό που θέλουμε είναι τουλάχιστον να επιβάλλουμε την ε, τήρηση και τη συμμόρφωση προς το ISO 26000. Ε, Ιδίω για τις εταιρείες που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο και για τις ανώνυμες εταιρείες, ώστε να τις υποχρεώσουμε να τηρούν αυτές τις δεσμεύσεις. Έτσι ώστε να μην ε, απαιτούμε μόνο την ε, δημοσίευση των ισολογισμών των εταιριών αυτών, αλλά και τα στοιχεία της κοινωνικής ευθύνης. Έτσι ώστε να υποχρεωθούν οι εταιρείες αυτές να ενσωματώσουν ε, στις επιχειρηματικές τους ενέργειες ε, την κοινωνική ευθύνη. Έχουμε βεβαίως τις διμερείς ε, συμφωνίες όπου σε πολλούς τομείς έχει σαχθεί αυτή η πτυχή της κοινωνικής ευθύνης. Αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε και περαιτέρω και να απαιτήσουμε μεγαλύτερη δέσμευση για να μπορέσει το θέμα της κοινωνικής ευθύνης να προαχθεί και να γίνει σεβαστό ε, μέσω των ευρωπαϊκών εταιριών και σε άλλα μέρη του κόσμου. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Ε, η Ελβετία, η οποία δραστηριοποιείται με διάφορες επιχειρήσεις στην Κολομβία, έχει συνάψει μια συμφωνία όπου οι ελβετικές εταιρείες υποχρεώνονται να, ε, σε, σεβαστούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις δραστηριότητες τους στην Κολομβία και γι' αυτό θα χρειαστεί οπωσδήποτε να συζητήσουμε περαιτέρω την εισαγωγή του στοιχείου της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την ενίσχυσή του στις εμπορικές μας συμφωνίες. Και τρίτον, η εταιρική κοινωνική ευθύνη σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τα προϊόντα τα οποία παράγονται. Όταν δείτε το iPhone σήμερα και το χρησιμοποιείτε και όταν πληρώνεις πολλά λεφτά στον, την Αμερικανική εταιρεία που τα κατασκευάζει. Θα πρέπει, νομίζω, είναι σωστό να ρωτήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες ε, κατασκευής του iPhone διεθνώς. Και άμα εξετάσουμε έτσι λεπτομερώς τις συνθήκες παραγωγής, θα δούμε ότι σε πολλά σημεία της παραγωγής δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις ε, που πρέπει της κοινωνικής ευθύνης. Και γι' αυτό ενδέχεται να μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε μία ετικέτα ε, κοινωνικής ευθύνης όπως έχουμε κάνει και άλλες ετικέτες, οι οποίες θα δείχνει ότι η εταιρεία αυτή συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες οδηγίες και υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να μετατοπίσουμε τον άξονα από την, από την εθελοντική συμμετοχή στη δεσμευτική συμμετοχή και υιοθέτηση των κανόνων αυτών και να μείνουμε στον σεβασμό αυτό, αυτής της ε, έννοιας της κοινωνικής ευθύνης σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική εισαγωγή της παρουσίας σας. Ανοίγουμε τη συζήτηση. Φρανσίς Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και την παρουσίαση των απόψεών σας με τις οποίες συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό. Δεν, χρειάζεται, δεν μπορούμε να έχουμε εθελοντικά πράγματα. Χρειαζόμαστε δεσμευτικές διατάξεις και πρέπει να μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσει Και η πρόταση της Κομισιόν δεν πάει προς τα εκεί που θα θέλαμε δεν είναι επαρκής ε, η συνένεση για να τηρούν τις υποσχέσεις τους οι επιχειρήσεις. Στο παρελθόν, για παράδειγμα, παρατηρήσαμε ότι τα εθελοντικά συστήματα όπως υπάρχουν δεν ήταν παρά μια βιτρίνα. Για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η Daimler, η BMW συμμετείχαν σε, αυτό το παγκόσμιο, σε αυτή την παγκόσμια σύμβαση, αλλά έχουν κάνει ελάχιστα για να μειώσουν τη ρήπανση ή, να, την, προστασία, για να, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρξε μια νέα μελέτη από έναν οργανισμό που αναφέρει τα προβλήματα σε αυτή την περίπτωση η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που δεν προλαμβάνει την εκμετάλλευση ανηλίκων. Μιλάμε για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τεράστια ρήπανση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα εθελοντικά συστήματα δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν καθόλου. Αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι δεσμευτικές διατάξεις. Χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε κυρώσει. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω και την Κομισιόν κατά πόσο διατίθεται να πάει πέραν των εθελοντικών συστημάτων. Αν όχι, Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποφύγουμε τις παραβιάσεις τους με άλλο τρόπο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο τρόπο από τις δεσμευτικές διατάξεις. Βλέπουμε ότι και σε άλλους τομείς δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα με τις εθελοντικές κατευθυντήρες γραμμές. Ποια είναι η στρατηγική σας λοιπόν για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την πρόληψη της ε, τη της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πολ Μέρφυ. Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας. Πιστεύω ότι στην φάση έχουμε 20 ετή εμπειρία από είχαμε πολλές ε, περιβαλλοντικές ε, καταστροφές που προκλήθηκαν από διαφορές επιχειρήσεις καθώς και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το συμπέρασμα που συναγούμε ότι και συμφωνούμε όλοι σε αυτό ότι αν αυτά τα πράγματα παραμένουν εθελοντικά, ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό δεν αξίζει το χάρτη που χρειαζόμαστε για να τα τυπώσουμε. Χρειαζόμαστε δεσμευτικέ διατάξει ορισμένε από τι επιχειρήσει ε, πολύ υψηλού προφίλ ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη παραβιάζουν οι ίδιε ε, βασικά κοινωνικά δικαιώματα και βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Έχω μια πολύ όμορφη έγχρωμη έκθεση της ΣΕΛ για την ε, εταιρική κοινωνική της ευθύνη που αποτελεί εξαιρετικό παραδείγμα greenwashing. Προέρχεται από... Γνωρίζουμε τι έχει γίνει με τους ακτιβιστές στην Ιγυρία, αλλά ουσιαστικά έχουν ε, αρπακτικές τεχνικές σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνεχίζουν και συνεχίζουν και στην Ευρώπη και στη Δυτική Ιρλανδία η Coca-Cola, άλλη μια εταιρεία που έχει μια εξέχουσα πολιτική CSR, συνεχίζει και πάλι να καταστρέφει τους υδάτινους πόρους, ειδικότερα στην Ινδία, εις βάρος του τοπικού πληθυσμού, η BP φυσικά, η British Petroleum, πολλά πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων, όπως αναγνωρίζει η Κομισιόν στο έγγραφο, χρησιμοποιούν τη CSR ως ε, τακτική που ουσιαστικά τη χρησιμοποιούν για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Ο Μίλτον Φρίντμαν είχε πει κάτι ωραίο ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι να κάνει μια επιχείρηση κέρδη. Δεν συμφωνώ, αλλά ουσιαστικά με τον τρόπο που είναι δομημένη η οικονομία μας και η επιχείρηση μας, αυτή είναι η πραγματικότητα αν δεν έχουμε δεσμευτικούς κανονισμούς ε, που να απαγορεύουν στις επιχειρήσεις κάτι τέτοιο, ουσιαστικά μεγιστοποιούν τα κέρδη τους εις βάρος ε, οποιοδήποτε άλλου θέματος. Και αυτό που, με, που αναρωτιέμαι για το έγγραφο της Κομισιόν που ήδη δεν είναι αρκετά δεσμευτικό, ουσιαστικά καταδικάζει τις εταιρείες που κάνουν, πραγματοποιούν greenwashing, αλλά από μια άποψη ουσιαστικά επιχειρεί greenwashing σε όλη την Ευρώπη μιλάει για χρήση της USR, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Υπάρχει απουσία εμπιστοσύνης ε, στις επιχειρήσεις και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιχειρησιακή εταιρική ευθύνη, την ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη για να καλυτερέψουμε τη φύση των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά αυτό που χρησιμοποιούν εταιρείε σε τοπικό επίπεδο προσπαθούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ευρύτερο επίπεδο. Χρειαζόμαστε δεσμευτικές διατάξεις και χρειαζόμαστε οι εταιρείε να είναι υπόλογες προς τους ανθρώπους. Ο Παβελ Ζαλεύσκη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Χάζεκ που δεν κατάφερε να συμμετέχει και να παρευρίσκεται σε αυτή τη συζήτηση. Είχε ετοιμάσει κάποιες σκέψεις που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Τις ε, σε γραπτά, γι' αυτό θα τις διαβάσω. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ε, διακυβέρνησης ε, έχει επιδεινωθεί. Πολλές επιχείρησεις ενδιαφέρθηκαν και χρησιμοποίησαν την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Συνεπώς ε, φαίνεται εμφανές ότι χωρίς την κατάλληλη προσέγγιση οι επιχειρήσεις στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν εμπόδια που θα είναι δύσκολο να υπερβούν. Σήμερα οι εταιρείε αντιλαμβάνονται το πλεονέκτημα της αηφορίας ως πηγή καινοτομία και δημιουργίας νέων επιχειρησιακών ευκαιριών. Όλοι αυτοί οι παράγοντε είναι κρίσιμη σημασία από πολλές ε, απόψεις. Το διεθνές εμπόριο δεν μπορεί να διεξάγεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο για τις διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις ε, είναι σημαντικό να επηρεάζουν θετικά τις κοινωνικές συνθήκες και την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να δοθεί λοιπόν πλήρης προσοχή στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σίγουρα η ανακοίνωση αυτή που αποσκοπεί στη δημιουργία συνθήκων ευνοϊκών για την αηφοροανάπτυξη, την υπεύθυνη επιχειρησιακή συμπεριφορά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να είναι ευπρόσδεκτο ως ένα ρεαλιστικό έγγραφο, ωστόσο πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να το βελτιώσουμε, να τη βελτιώσουμε ώστε η πολιτική ιατρική κοινωνική ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια, ένα σύγχρονο καινοτόμο εργαλείο που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τι τρέχουσε προκλήσει που θέτει το εμπόριο όπω είναι σήμερα διεθνώ. Συντάσσοντα τη σχετική γνωμοδότηση υπάρχουν πολλά ζητήματα στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε όπω η βελτίωση των ε, ηθικών συμπεριφορών των επιχειρήσεων σε σχέση με το διεθνέ εμπόριο, να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις, να υλοποιήσουν κώδικες διοντολογία που να συμμορφώνονται με τις αρχές εταιρική κοινωνικής ευθύνης, μείωση της γραφειοκρατίας και οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών σε σχέση με θέματα εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ε, όσον αφορά την άποψη του Συμβουλίου η προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας είναι σημαντική και πρέπει να τονίσουμε ότι από την άψη της δικής μας Επιτροπής είναι σημαντικό να εισάγουμε κανονισμούς που θα διασφαλίζουν ότι το διεθνές εμπόριο θα είναι υπεύθυνο κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Πιστεύει λοιπόν η συνάδελφος ότι η πρόκληση δημιουργίας μιας νέας στρατηγικής σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί κρίσιμο βήμα για τον επανασχεδιασμό του αποτελέσματος του CSR. Το ζήτημα δεν είναι κατά πόσο συμπεριφέρεται κοινωνικά υπεύθυνα μια επιχείρηση, αλλά μάλλον το πόσο αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά. Οι υπεύθυνε επιχειρήσει εξαρτώνται από εμά. Η κυρία Χάντσεκ πιστεύει ότι η επικοδομητική συζήτηση και η στενή συνεργασία θα μπορέσουν να παράσχουν μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ριβεμπέ τελικά, μέρος της ελιστικής ομάδας. Θα ήθελα και εγώ να παρουσιάσω εκ μέρους του Αρλέμ Τεζίν αυτές τις ιδέες. Ζητά συγγνώμη που είναι απόν αυτή τη στιγμή προεδρεύει του ε, Προεδρείου της Σοσιαλιστικής Ομάδας στη Γαλλία. Δεν θα γίνει πρώτος γραμματέας, αλλά γενικός γραμματέας, αλλά πρώτος γραμματέας της Σοσιαλιστικής Ομάδας στη Γαλλία. Χαιρετίζω το γεγονός ότι είναι έμπειρος ευρωβουλευτής, ε, τρεις θητείες έχει κάνει, ήταν και πρόεδρος σοσιαλιστικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, Αρλέμ, μέλος πολύ ενεργό αυτής της Επιτροπής και όπως ξέρετε είναι ανοιχτό στην ευρωπαϊκή προβληματική. Δεν έχει παροπίδες και δεν βλέπει μόνο τη Γαλλία Βλέπει όλη την Ευρώπη μπροστά του και βεβαίως του είναι ιδιαίτερα προσφυλής όλοι αυτοί οι κανόνες για να μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, να εφαρμόσουμε κάποιες ιδέες και να ακολουθήσουμε κάποιες κοινέ. Και τώρα καλείται να γίνει πρώτος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος στη Γαλλία. Τώρα, για το θέμα αυτό το οποίο τον απασχόλησε δεν θα πω τώρα σε λεπτομέρειες των δικών του προτάσεων. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μιλούμε στον παρατατικό, διότι ούτω ή άλλως θα παραμείνει ευρωβουλευτής ο Αγλέμ ε, Ντεζίρ. Ίσως θα είναι λιγότερο διαθέσιμο από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά παρόλα αυτά θα παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλο αυτή τη Επιτροπή μα. Θα συμμετέχει λοιπόν και στο μέλλον ε, στην ε, εργασίες μας και θα εμπλουτίσει το κείμενο το οποίο σας παρουσίασε και ο Μπερτ Λάγκε. Το πρόβλημα είναι ποιος είναι, σε ποιο ποσοστό θα μπορέσει το θέμα αυτό να καταστεί υποχρεωτικό. Ένα μόνο. Ποιος είναι όμως αυτός ο οποίος παίρνει αποφάσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα. Ο ΠΟΕ, Διεθνής Οργανισμός ε, Εμπορίου, έχει το σχετικό ε, δικαστήριο πρωτοδικείο στο οποίο μπορεί κανείς ε, να απευθυνθεί, να προσφύγει εάν υπάρξει παραβίαση επιβάλλει πολύ σημαντικά πρόστιμα αλλά όλοι οι υπόλοιποι η Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, η Διεθνής Οργάνωση Υγείας, το ΠΝΙΔ, όλες οι άλλες μεγάλες διεθνεί οργανώσει που ανήκουν στην οικογένεια του ΟΗΕ εκφράζουν επιθυμίες πολιτικού, ηθικού χαρακτήρα, αλλά είναι προαιρετικές, δεν είναι υποχρεωτικές. Θα ήταν ένα μεγάλο βήμα προόδου της του πολιτισμού και θα φτάσουμε σε πολύ καλύτερο σημείο ισορροπίας των πραγμάτων αν μπορέσουμε να κάνουμε κάπως υποχρεωτική την ε, υποχρέωση τήρησης των διεθνών κανόνων και προδιαγραφών. Στα πλαίσια της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας δεν προβλέπεται να ακολουθούν όλους τους κανόνες της, ε, τους ε, κοινωνικούς που ισχύουν είτε στη Σουηδία ούτε στην ε, Ελβετία. Έχει όμως θεσπίσει οκτώ θεμελιώδους σημασίας και απλούς κανόνες. Δηλαδή τα παιδιά πάνε στο σχολείο, δεν δουλεύουν στα εργοστάσια. Οι μισθωτοί έχουν το δικαίωμα να οργανωθούν συλλογικά για να διαπραγματευτούν την σύμβαση της λογική τους. Δεν πρόκειται εδώ για κανόνες των πολσεβίκων, αλλά για βασικούς κανόνες. Το να κάνουμε λοιπόν υποχρεωτικού αυτού του υποχρεωτικού βασικού κανόνε, πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα γιγαντίο βήμα προ τα μπρο. Και θα πρέπει να σκεφτούμε και ένα άλλο θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από νομική πλευράς να καταστήσουμε υπεύθυνε τι μεγάλες πολυεθνικές και τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ε, έδρα ή θυγατρικές στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα πρέπει η διεύθυνση αυτών των επιχειρήσεων να καταστούν υπεύθυνε των πράξεών τους και του τρόπου με τον οποίο ενεργούν. Διότι σήμερα, επειδή δεν είναι υποχρεωτικό ότι κάτι τέτοιο, ότι φλούν, στρέφουν αλλού το βλέμμα και αν υπάρξει νομικό πλαίσιο, αν μπορέσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο που θα τις καταστήσει υπεύθυνε, ώστε τα θύματα των κοινωνικών περιβαλλοντικών καταστροφών να μπορούν να προσφύγουν σε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουμε κατορθώσει κάτι. Ξέρουμε ποιο είναι το σύστημα ε, που βασίζεται στην εθελούσια μας. Πρέπει να πω ότι από τις ε, χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ευρώπη, μόνο λίγες είναι αυτές οι οποίες κάνουν ε, εκθέσεις που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το υποχρεωτικό χαρακτήρα να τον ενισχύσουμε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Ξέρω ότι είναι πιο εύκολο να κάνει κανεί κάτι παρά να ενεργεί. Τα λόγια είναι πάντα πιο εύκολα από τα έργα, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Μεκρή, με, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ορί ε, και καλά έκανες και υπογράμμισες το ρόλο του ε, Αγλέμ Ντεζίρ στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα και εγώ ως πρόεδρος και προσωπικά να συγχαρώ το Σοσιαλιστικό Γαλλικό Κόμμα που εξέλεξε ως πρώτο γραμματέα ένα αξιότιμο μέλος της δικής μας Επιτροπής. Και χαίρομαι που άκουσα ότι θα συνεχίσει να είναι μέλος της Επιτροπή μας. Διερωτώ με, μπορεί κάποια άλλη Επιτροπή να είναι τόσο υπερήφανη, διότι μεταξύ των μελών της αριθμοί και έναν τόσο σημαντικό πρωτογραμματέα κόμματος, μια τόσο σημαντική χώρα. Ο κύριος Τόμας Ντότ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, χαίρετε. Σύντομα, για αυτή τη νέα έννοια και αντίληψη αυτής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πρόκειται για την ευθύνη των εταιριών για τις επιπτώσεις των πράξεών τους και των δράσεών τους στην κοινωνία. Οι επιπτώσεις αυτές, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πρέπει να το πούμε ότι είναι συνήθως θετικές, αλλά μπορεί ενίοτε να είναι και αρνητικές. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να εργαστούμε και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις. Η πολιτική μας είναι αυτή, να γίνει αυτό με ισορροπημένο τρόπο. Δηλαδή, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν τα θετικά που κάνουν και να εντοπίσουμε και να αμβλύνουμε και να προλάβουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των δράσεών τους. Ο ορισμός λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικός διότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν επίπτωση στο περιβάλλον που ρεύουν. Συνήθως θετικό, αλλά πολλές φορές αρνητικό επίσης. Όλοι το κάνουν αυτό. Άρα όλες οι επιχειρήσεις έχουν κοινωνική ευθύνη. Και τα μέλη της Επιτροπής σας θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο λέγεται είναι εθελοντικό, είναι υποχρεωτικό. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να υπάρχει τέτοιου είδου κοινωνική ευθύνη. Το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να περιμένουμε να ανταποκριθούν σε αυτή την κοινωνική ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εμείς πρώτα απ' όλα τι λέμε, πρέπει να συμμορφούνται με τους νόμους και δεύτερον να ενσωματώνουν κάποια θέματα στην πολιτική τους και τη στρατηγική τους σύμφωνα με τα ε, εμπλεκόμενους σε λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, την τήρησή τους, τα θέματα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά. Υπάρχουν ε, πρώτα απ' όλα οι εταιρείε, οι πολυεθνικές, οι οποίες πρέπει να ε, τηρούν κάποιες διεθνείς συμφωνίες, κάποιους κανόνες, να τους ασπάζονται και τους ακολουθούν η πολιτική μας, η συνεταιρική κοινωνική ευθύνη κάνει κάτι καινούριο. Δεδομένου ότι αναγνωρίζει πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει μια συμπληρωματική νομοθεσία. Πράγμα που δεν είναι, που είναι κάτι καινούριο. Και βεβαίως αυτό ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα, δεδομένου ότι έχουμε την κατάλληλη εθνική και κοινοτική νομοθεσία για να πληρούνται αυτή η κοινωνική εταιρική ε, ευθύνη και θα πρέπει απλώς αφού αναγνωριστεί κάτι τέτοιο να γίνει και πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει στο μανίκι της ένα άσο η Επιτροπή για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική και προσπαθεί να την προτείνει ώστε να αποτελέσει μέρος της κοινωτικής νομοθεσίας. Η δέσμευσή μας είναι επίσης ε, να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις προφορίες μη ε, ε, οικονομικού χαρακτήρα σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να επιβάλλουμε κάποιες ειδικές δραστηριότητες σε κάποιες επιχειρήσεις, διότι ζητούν ε, Φερρυπίν στην Γαλλία και στην Δανία ζητάει η νομοθεσία να αποκαλύπτουν κάποιες από τις δραστηριότητες τους. Και αυτό είναι μέρος δικής νομοθεσίας. Τώρα, όσον αφορά αυτό το ε, ε, εθελοντικό χαρακτήρα, αν κάτι τέτοιο έχει κάποια ισχύ ή όχι, κυρίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είμαστε τόσο απεσιόδεξοι όσο κάποιοι συναδελφοί σας που εξέφρασαν απόψεις για τον ε, χαρακτήρα αυτών των ε, πρωτοβουλίων σε, εθελοντικό, σε εθελοντική βάση ή σε νομικά υποχρεωτική βάση. Ξέρουμε ότι σε διάφορες ε, τομείς, σε διάφορες επιχειρήσεις ακολουθούνται κάποιες αρχές και για την πράσινη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ισχύουν και στον, στον ΟΗΕ. Πρόκειται για κάτι το σημαντικό, διότι εδώ δεν μιλούμε μόνο για επιχειρήσεις, αλλά για τις προσδοκίες του τι πρέπει να κάνουν οι διάφορες επιχειρήσεις για να μην ε, ε, δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πράγμα που σημαίνει ότι και τα κράτη πρέπει να υπακούν σε αυτούς τους κανόνες. Βεβαίως δεν είναι κράτος η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό προσπαθήσαμε στην Επίτροπη να συντάξουμε μια έκθεση για να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις αρχές στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση, ας επιστρέψουμε στον ε, εισηγήτη μας, τον κύριο Λάγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι... Ε, α, μάλλον δεν με ικανοποίησε η παρέμβαση της Κομισιόν. Ε, εντάξει, διαγράφεται ένα νέο βήμα προς μια καινούργια κατεύθυνση, αλλά ε, εδώ πρέπει να εδραιώσουμε καινούργια μέτρα κατευθυντικές γραμμές και άλλα πιο ήπια μέτρα ε, πρέπει να είμαστε συνεπείς διότι εάν δείτε τον τομέα των εμπορικών συναλλαγών και τις άμεσες επενδύσεις σε άλλες χώρες, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία και ε, πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζουν και την κοινοτική νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε άλλες απαιτήσεις στις δικές μας ευρωπαϊκές εταιρείες. Γι' αυτό ε, πρέπει να τις πείσουμε εκτός από τον σεβασμό των κανόνων του διεθνούς εμπορίου να υλοποιήσουν και διεθνείς προδιαγραφές, σαφείς προδιαγραφές, σαφείς κανόνες για την εφαρμογή του, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και ε, πρέπει γι' αυτό να έχουμε εμείς προδιαγραφές και κανόνες τις οποίες να μπορούν να ακολουθήσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Αυτά είναι θέματα τα οποία σίγουρα θα συνεχίσουμε να συζητάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη ε, το επόμενο βήμα αυτού του φακέλου είναι να το συζητήσουμε στις 6 Νοεμβρίου. 6 Νοεμβρίου όπου θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης η οποία θα, την οποία θα παρουσιάσει ο εισηγητής. Τώρα, κοινή συζήτηση, ε, σημεία 29-30, για την εφαρμογή των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ε, συμπλήρωση του παραρτήματος του κανονισμού Αυτό για διασμολογική και στατιστική ονοματολογία και του κοινού δασμολογίου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Βραζιλία, Ταϊλάνδη. Και ε, την ε, νομοθεσία γενικά η οποία χρειάζεται για την τραποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο πολιτικών μεταξύ των χωρών αυτών που ανέφερα. Φέτος τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τις συμφωνίες με τη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη για την τραποποίηση των παραχωρήσεων σε αυτά τα δύο προϊόντα με τα κρέας και πουλερικά. Ο λόγος αυτής της τροποποίησης είναι ότι οι εισαγωγές ε, μεταποιημένου κρέατο και πουλερικών στην ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκαν γεωμετρικά. Και λόγω της εκμετάλλευσης ορισμένων ε, ασαφών ε, σημείων ε, της συμφωνίας που υπήρχε. Έτσι λοιπόν εκμεταλλεύτηκαν ορισμένα συγκεχημένα σημεία, ορισμένες ασαφείς διατάξεις και μπόρεσαν να αυξήσουν αστρονομικά τις εισαγωγές τους και έπρεπε να υπάρξει μια αντιστάσμιση αυτής της κατάστασης. Και για να αντισταθμίσουμε τα συμφέροντα των εμπορικών μας εταίρων, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ε, επιτρέψει ορισμένες ποσοστώσεις στις χώρες αυτές και γι' αυτό χρειάζεται η τροποποίηση αυτή. Ε, προσπαθούμε με αυτές τις τροποποίησεις να διορθώσουμε ένα σφάλμα ένα σφάλμα που σημειώθηκε σε αυτή τη συμφωνία σχετικά με τις εισαγωγές αυτού του είδους μεταποιημένου κρέατος. Γι' αυτό η σύστασή μου είναι να συμφωνήσουμε, να, να δεχθούμε αυτή τη συμφωνία. Και θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις των μελών της Επιτροπής μας για αυτά τα δύο θέματα, εάν υπάρχουν απόψεις. Ε, ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο από αυτά που είπατε εσείς. Ε, κάνατε μια πολύ καλή και περιεκτική σύνοψη μιας περίπλοκης κατάστασης και ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας. Αυτά είχα να πω εκ μέρους Κομισιόν πριν μικρά λαθάκια να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Ωραία, δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις στη σύστασή μου. Αλλά η προθεσμία των τροπολογιών στο σχέδιο έκθεσης και στο σχέδιο σύστασης είναι 20 Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας τον Οκτώβριο. σφοφορία τον Οκτώβριο, προθεσμία των τροπολογιών 20 Σεπτεμβρίου. Και προχωρούμε στο τελευταίο θέμα ε, της σημερινής ατζέντα 31. Και φτάνουμε στο τέλος αυτής της μακράς συνεδρίασης 31. Είναι το ένα ε, σημείο, το εκρεμές σημείο του φακέλου για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Ο ίδιος εισηγητής είναι όπως και πριν και πάλι είναι μια γνωμοδότηση για την εσωτερική αγορά, η οποία είναι επί της ουσίας η και εμείς ε, συντάσσουμε τη γνωμοδότηση. Ας ακούσουμε λοιπόν τον εισηγητή. Τζαν Λούκα Σούστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεδομένη τη πολλοπλικότητα του θέματο και ότι δεν, έχουμε διαθέσιμο το κείμενο, δεν είχαμε διαθέσιμο το κείμενο του κυρίου Συγητή το Ζουβά τον Ιούλιο, χρειαστήκαμε περισσότερο χρόνο για να σκεφτούμε αυτή την πρόταση οδηγία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο και λόγω κάποιων πολύπλοκων θεμάτων που προήλθαν από την ε, κύρια θα έλεγα Επιτροπή για την ίδια την οδηγία της ΣΥΜΚΟ θα ήθελα να αναδείξω την... πόσο ωφέλιμη είναι αυτή η οδηγία την οποία ορισμένοι αμφισβητούν διότι μέχρι στιγμής οι διατάξεις για το θέμα των παραχωρήσεων έχουν διαμορφωθεί κυρίως για να μην πω αποκλειστικά από τη δικαιοδοσία και τους εθνικούς κανόνες αντί για τις ε, γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, μια κανονιστική παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει δεκτή για ένα νομικό πλαίσιο πιο καθαρό θα έχει όφελος και για, τους διεθνείς, ε, για τις διεθνείς επιχειρήσεις. Επίσης ε, είναι ανάγκη να μελετήσουμε προσεκτικά το έργο του συναδέλφου κ. Ζουβά που περιλαμβάνει κατευθύνσεις θετικές για την αναδιοργάνωση του κειμένου που προτείνει η Εκτελεστική Επιτροπή. Θα έλεγα ότι σήμερα που γνωρίζουμε το κείμενο μιλάμε για πολύ δυσδυτικές ε, τροποποιήσεις που θα μπορέσουν να επιλύσουν τα πιο ακαθόδη ζητήματα αυτού του προβλήματος. Είμαστε λοιπόν υπέρ τη αναδιοργάνωση, της απλούστευση της αυτονομίας των εθνικών αρχών σε αυτόν τον τομέα, καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας και των διαδικασικών ανάθεσης έργων, χωρίς να χάνουμε τις βασικές αρχές σε ένα τόσο σημαντικό τομέα όσο των συμβόσεων παραχώρησης και τον έλεγχο της νομιμότητα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβουμε δραστικά στα ζητήματα προσαρμογής των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών ζητημάτων, στα δικαιώματα των εργαζομένων ε, μέσα στα κριτήρια ανάθεσης καθώς και την αξιολόγηση των υποψηφίων, τα κριτήρια αποκλεισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουμε ήδη κάνει στην οδηγία για τις δημοσίες συμβάσεις και για τις υπηρεσίες κοινής οφειλίας. Θεωρώ επίσης ότι καλό είναι να περιορίσουμε το κριτήριο ανάθεσης των παραχωρήσεων στο άρθρο 39 της πρότασης οδηγίας βάσει μια σειράς κριτηρίων που θα ε, δοθούν στις διοικήσεις που θα αναθέτουν τα έργα. Καθώς και η εξέταση του κόστους του κύκλου ζωής του διαγωνισμού είναι σημαντικό να εισάγουμε μια διάταξη δεσμευτική που θα σχετίζεται με τις ε, τυχόν προσφορές τρίτων χωρών. Με σκοπό επίσης να υπάρχει επίπεδο αμοιβαιότητας μεταξύ στην ευρωπαϊκή αγορά όπως και στις τρίτες χώρες προσέχοντας να κάνουμε διάκριση μεταξύ των ανεπτυγμένων και των πιο φτωχών χωρών. θεωρώ ότι πρέπει να χαμηλώσει το κατοφλείο των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ε, Αγαπητέ συνάδελφε, πηγαίνετε πολύ γρήγορα και λυπάμαι οι διερμηνείς. Ε, μπορείτε να μιλάτε λίγα λιγάκι πιο αργά, παρακαλώ. Και στο θέμα των παραχωρήσεων, ε, που έχουν συμπεριληφθεί στις οδηγίες για τις δημοσίες συμβάσεις και για τις ε, υπηρεσίες κοινής ωφελίας, στο σχέδιο γνωμοδότης επίσης σκέφτηκα να προτείνω τη μείωση του κατοφλίου για τις παραχωρήσεις υπηρεσιών από 5 εκατομμύρια ευρώ σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και θεωρώ ότι όλοι θα συμφωνήσουν με την ιδέα του εισηγητή κ. Ζουδά να χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης το τιμολόγιο που ε, έχει εκτιμήσει ο παραχωρών θα πρέπει να τηρήσουμε την αρχή της εφαρμοσιμότητας της οδηγίας μόνο σε μελλοντικέ παραχωρήσεις και να μην έχει εφαρμογή στις τρέχουσες συμβάσεις, ώστε να μην έχουμε δικαστικά προβλήματα μεγάλης ευρύτητας ε, όταν θα ανοίξουν οι αγορές σε αυτό το σύστημα επιλογής Διαφορετικά, αν θέλουμε να τροποποιήσουμε τις τρέχουσες συμβάσεις, θα πρέπει να εισάγουμε συγκεκριμένα κριτήρια. Στο σύνολο μου φαίνεται εξαιρετικό το έργο, αλλά έχουμε ακόμα μια εβδομάδα ώστε να εργαστούμε και να μπορέσουμε να παράγουμε τις τροπολογίες εκείνες που θα προσαρμόσουν την πρόταση περισσότερο στις προθέσεις του Κοινοβουλίου και στην ομολογία που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησή σας που έχετε στο αρχείο σας. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Δεν βλέπω να υπάρχουν ε, παρατηρήσεις. Ας ακούσουμε την Κομισιό, την κυρία Σίσοφκα. Συγγνώμη, λέει πρόεδρε, δεν μπορώ να προφέρω σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την έκθεση γνωμοδότησης και για την αναγνώριση ότι θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες για το θέμα των παραχωρήσεων. Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι ο στόχος αυτής της οδηγίας είναι αφενό να εγγυηθεί διαφάνεια, ή μεταχείριση, έλλειψη διακρίσεων μεταξύ των οικονομικών φορέων, αλλά και νομική ασφάλεια στο δημόσιο, ώστε να γνωρίζουν ότι οτιδήποτε σύμβαση γίνει υπό αυτού του όρου δεν θα έχει νομικά κενά. αναφέρθηκε το πλαίσιο για τον ορισμό και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει αυτέ οι παραχωρήσει να ορθώνονται. Επίση, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσει σε σχέση με αυτά που εισηγηθεί. Δεδομένου ότι σήμερα δεν υπάρχουν καθόλου κανόνε και δεν υπάρχει νομική σαφήνεια για το τι ακριβώ πρέπει να λάβουμε υπόψη Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσταση τη Επιτροπή είναι πάρα πολύ σαφή. Και τα πράσινα και τα κοινωνικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στον τομέα των παραχωρήσεων. Και θα ήθελα σε μία από τις παρατηρήσεις που έκανε στο τέλος ο εισηγητής να πει ότι οτιδήποτε γίνει θα αφορά τις μελλοντικές ε, συμβάσεις παραχώρητες. Η διαδικασία μας είναι να συνεργαστούμε περαιτέρω μαζί σας ώστε να υπάρχουν ε, περαιτέρω διευκρινήσεις και να χτενίσουμε το κείμενο ώστε να βγει τέλειο το τέλος. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Τζανλούκα, θες να προσθέσεις κάτι. Σχόλια μετά από την... Σχόλια της Επιτροπής. Όχι. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχουν σχόλια, Η διαδικασία. 7 Νοεμβρίου ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 28 Σεπτεμβρίου. Και φτάσαμε στο τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Και από εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτε, ούτε κι εσείς. Η επόμενη συνεδρίαση 10 και 11 Οκτωβρίου Αρχίζουμε στις 10 το απόγευμα. Στις 3 ακριβώς παρακαλώ. Γιατί όλο και περισσότερο καθυστερούμε να αρχίσουμε. Παρακαλώ λοιπόν να είστε στην ώρα σας. Ευχαριστώ και χαιρετώ.